Ξεκινούμε την κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Γυναικών και Ισότητας ε, των Φύλων. Έχουμε κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών Γεωργίας και Γυναικών. Και αυτό γίνεται προκειμένου να ψηφίσουμε την έκθεση για τις γυναίκες και το ρόλο τους στις αγροτικές περιοχές. Οι συγκήτριες είναι η κυρία Μαριάννα Πετήρ και η κυρία Σένρα Ροντρίγκες περίμενα λίγο ε, και γι' αυτό καθυστέρησα να ξεκινήσω τη συνεδρίαση γιατί βλέπω ότι ακόμη υπογράφουν ε, μερικοί ευρωβουλευτές. Οπότε τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλωσορίζω εγκάρδια κυρίως ε, τους ευρωβουλευτές από την Επιτροπή Γυναικών. Έχουμε εδώ και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Γυναικών. Ε, είναι ο κύριος Πιμέντα Λόπες, ε, που θα του δώσω το λόγο για λίγο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ε, ευγένειά σας και την καλοσύνη που είχατε να μου δώσετε το λόγο. Δεν πρόκειται να μακρηγορήσω. Θα ήθελα εκ μέρους Επιτροπής Γυναικών και Ισότητας των Φίλων να εκφράσω τις ευχαριστίες μου για την αγαστή συνεργασία που είχαν οι δύο επιτροπές μας και να επενέσω τις εισηγήτριες ε, για την προσπάθειά τους και τη συνεργασία τους με τους και εισηγητέ. Κατάφεραν να καταλήξουν στις συμβαστικές προτάσεις ώστε να καταρτήσουμε ένα ισορροπημένο έγγραφο για το ρόλο και τη συμβολή των γυναικών στις αγροτικές περιοχές αφενός και αφετέρου να εξασφαλίσουμε ένα δρόμο, μια σωστή κατεύθυνση και να ξεπεράσουμε τις ανισότητες μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα αυτό. Αυτά, όπως σας υποσχέθηκα, ήμουν λακωνικός και θα δώσω και πάλι το λόγο στον Πρόεδρο για να περάσουμε στην ψηφοφορία. Σας ευχαριστούμε κύριε Λόπες. Θέλει μήπως κάποια από τις να λάβει το λόγο. κάποιος ε, ίσως από τους καλούς συγκεκριτές. Κύριε Πετήρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους. Όλους τους συναδέλφους που με τις προτάσεις τους, τις τροπολογίες τους ε, και τη συμβολή τους ε, απέδειξαν ε, πόσο σημαντικό είναι για όλους μας ε, να αναβαθμίσουμε το ρόλο των γυναικών στις αγροτικές περιοχές. Θεωρώ ότι η έκθεση που εκπονήσαμε είναι πολύ θετική και θα καταφέρουμε να την εγκρίνουμε στη σημερινή ψηφοφορία. Πρώτα απ' όλα όμως θα ήθελα να πω ότι αφιερώνω αυτή την έκθεση σε όλες αυτές τις γενναίες, θαραλές Γυναίκε που μένουν στι αγροτικέ περιοχέ που μένουν στην Ήπεθρο, γιατί με το λειτουργικό του ρόλο διαφυλάσσουν την οικογένεια, την κουλτούρα μα, τι παραδόσεις μα, την πολιτιστική μα κληρονομιά, την βιοπικιλότητα, παράγουν και τρόφιμα, μας ασιτίζουν Είναι πραγματικές ηρωίδες οι γυναίκες στην Ήπεθρο και ελπίζω χάρη σε αυτή την έκθεση να αναβαθμίσουμε κάπως ε, το ρόλο τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Σένερα. Eh, Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη και εγώ να σας ευχαριστήσω και να ευχαριστήσω όσους ε, συνεισέφεραν στην ε, έκθεση αυτή και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις πολλές προσθήκες που έγιναν από τις διάφορες τροπολογίες και οι οποίες μας διευκόλυναν στο να καταθέσουμε σήμερα μια έκθεση αυτής της μορφής. Θα ήθελα επίσης να χρησιμοποιηθεί η έκθεση για να συνεχίσουμε με τις προσπάθειες που κάνουμε για να βελτιώσουμε και τις συνθήκες διαβίωσης αλλά και ε, στην εξασφάλιση των ίσων δικαιωμάτων σε όλες τις γυναίκες που ζουν στην Ήπεθρο. Ευχαριστώ. Ζήτησε το λόγο και η κυρία Μορβάη. Παρακαλώ. Ε, do I understand... Έχω καταλάβει σωστά πως γίνεται συζήτηση για την έκθεση ή δεν γίνεται συζήτηση, απλώς ψηφοφορία. Με συγχωρείτε. Όχι, όχι, μόνο ψηφοφορία, όχι συζήτηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω και τους καλεσμένους της κυρίας Πετήρ γυναίκες ε, από την Ήπεθρο, από τις αγροτικές περιοχές, ε, ήρθαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά από πρόσκληση της κυρίας Πετήρ. Σας ε, καλωσορίζω θερμότατα. Παίρναμε τώρα στην ψηφοφορία. Όπως προβλέπει η διαδικασία, τις συμβαστικές τροπολογίες θα τις ψηφίσουμε ηλεκτρονικά και θα δούμε αν συμφωνείτε να επιταχύνουμε την ψηφοφορία, να μην ρωτάω ε, κάθε φορά και τις ψήφους κατά και τις αποχές, αν βλέπω ότι η ψήφη υπέρ είναι πλειοψηφία. Ψηφίζουμε την ε, συμβαστική τροπολογία. 15 αρχίζουμε με ηλεκτρονικό τρόπο παρακαλώ. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται. Περνάμε στην 176. Ποιος είναι υπέρ παρακαλώ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 176. Ευχαριστώ. Κατά. Παρακαλώ. Ποιος θέλει το λόγο. Α, όχι, είπατε ότι η κάρτα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σας δεν λειτουργεί. Καλά, αλλά τα χέρια σας. Αλλιώ θα πρέπει να ελέγχουμε ηλεκτρονικά κάθε φορά το αποτέλεσμα. Λοιπόν, ποιο είναι υπέρ τη τροπολογία 176. Κατά. Απορρίπτεται. Δεν έχουμε αγγλική διερμηνία. Μια στιγμή παρακαλώ. Now Εντάξει τώρα. Εντάξει. Ψηφίζουμε την συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικό έλεγχο προηγουμένων όμω για την τροπολογία 176. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικό έλεγχο για την 176. Τέλο ψηφοφορία απορρίπτεται. Αλλά είχατε δίκιο γιατί ήταν οριακή διαφορά, οπότε καλό ο έλεγχος. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία συμβιβαστική 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 161, ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 161, παρακαλώ, κατά, απορρίπτεται. 144, ποιος είναι υπέρ, τροπολογία 144, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 144, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τη συμβαστική τροπολογία 18. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 306. Ποιος είναι υπέρ της 306. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 306. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Πρέπει να γίνει ηλεκτρονικός... Όχι, συγγνώμη. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 19. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ο κύριο Ταραμπέλα. Αναρωτιέμαι γιατί δεν ε, ψηφίσαμε την 174. Ε, δεν καταλαβαίνω. Είναι η κυρία Σάιερ Πύρικ. Γιατί δεν έχουμε ψηφίσει αυτήν. Σα ευχαριστούμε. Δικό μου λάθο, δικό μου λάθος, μέα ε, κούλπα. Καλά που μα το επισημάνατε. Τροπολογία 174. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα περνάμε. Η τροπολογία συμβαστική 19 έχει εγκριθεί. Αλλά σε επαναλάβουμε την ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 19, επανάληψη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ευχαριστώ. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε Στην τροπολογία 199. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 199. 199. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 200. Ποιος είναι υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 200 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται, αλλά με μικρή διαφορά, γι' αυτό έκανα και τον έλεγχο. Συμβαστική τροπολογία 20. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 21. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική τροπολογία 21. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 307. Ποιος είναι υπέρ της 307. Εγκρίνεται. Ευχαριστώ. Ποιος είναι υπέρ της 190. Τροπολογία 190. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 201. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 212. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 212 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 227. που είναι επανομοιότυπη με την 229. Θα ήθελα αν γίνεται να ελέξουμε την 190, γιατί νομίζω είπατε ότι απορρίπτεται και η δική μου εντύπωση είναι ότι έχει περάσει. Ναι, αλλά να αντιδράτε αμέσως στο μέλλον, να μην απομακρυνόμαστε τόσο από την τροπολογία. Εντάξει, αφού θέλετε, άρχεται ο ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 190. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Περνάμε στις τροπολογίες 227 και 229 που είναι πανομοιότυπες. Ποιος είναι υπέρ, κατά, ηλεκτρονικός έλεγχος, για τις δύο τροπολογίες, 227 και 229. Άρχεται η, τροπολογία, η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνονται, αλλά με μικρή διαφορά. Περνάμε στην ψηφοφορία της συμβαστικής τροπολογίας 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 244. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 172. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 251. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 24. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 297. Ποιος είναι υπέρ της 297? Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 243. Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 25. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία της συμβιβαστική 25. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 265 τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 245. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 246. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική τροπολογία 26. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 28. Άρχεται η ψηφοφορία για την συμβαστική τροπολογία 28. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 284. 284. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 284. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 284 Ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται οριακά, αλλά εγκρίνεται. Τροπολογία 309. Ή μήπως όχι. Όχι. Συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Όχι, διορθώνει ο πρόεδρος. Τροπολογία 309. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τώρα συμβαστική τροπολογία 27. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 294. Ποιος είναι υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της 294. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 300. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 300. Άρχεται η ψηφοφορία. 300. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 29. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 1 του κυρίου Μαριά. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 1 κατά Εγκρίνεται, αλλά ας το ελέγξουμε για καλό για κακό. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Zamykam ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 3. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 4. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 5. Ποιο είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 6. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 7. Υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην 127 της κυρίας Ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται, 127. Συμβιβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 105 της κυρίας Νταντσίλα. Ποιος είναι υπέρ της 105. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 58 της κυρίας Κρούπα. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 58. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 31. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβεβαστική τροπολογία 5. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 42 της κυρίας Μόη. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 42. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 51. Ποιος είναι υπέρ. Είναι της κυρίας Σέρα και λοιπόν, ποιος είναι υπέρ τη τροπολογία 51. Κατά. Απορρίπτεται, αλλά θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Για την τροπολογία 51. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ε, με μικρή διαφορά έπρεπε να γίνει έλεγχος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Ποιος είναι υπέρ της 34. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Περνάμε στην τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ της 60. Εγκρίνεται. Τροπολογία 61. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 65 υπέρ. Εγκρίνεται. 66 υπέρ. Εγκρίνεται. 68 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9 έρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τροπολογία 92. Ποιος είναι υπέρ της 92. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 73. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Περνάμε στην 126. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 126. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 22. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 106. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 106. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Με δύο ψήφους διαφορά έπρεπε να γίνει έλεγχος οπωσδήποτε. Τροπολογία 110. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεν σηκώνετε τα χέρια σας και πρέπει να κάνουμε έλεγχο. Άρχεται ε, ηλεκτρονικός έλεγχος για την 110. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 111 Ποιος είναι υπέρ? Εγκρίνεται. 112. Υπέρ. Α, λάθος. Γλωσσικό χωρίς ψήφο. Ε, συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική 13. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. εγκρίνεται. Έγιναν δεκτέ όλε οι βασικέ τροπολογίε. Ολοκληρώσαμε την ψηφοφορία και των υπόλοιπων τροπολογιών. Ψηφίζουμε το σύνολο ε, του ψηφίσματο όπω έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλο ψηφοφορία. Ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια στις ε, συνεισηγήτριες. και να σας ευχαριστήσω όλους για τη συνεργασία και την κοινή ψηφοφορία των δύο επιτροπών. Ευχαριστώ και τους βοηθούς και συγχαρητήρια και πάλι τις συνεισηγήτριες. Θέλει κανείς μήπως το λόγο? Όχι. Οπότε σας ευχαριστώ. Τρία λεπτά τεχνικό διάλειμμα για να σας αφήσουμε το χρόνο να φύγετε με βαριά καρδιά σας αφήνουμε να φύγετε, τα μέλη της Επιτροπής Γυναικών, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε κι εμείς. Νομίζω ότι τα καταφέραμε πάντω, κυρίες και κύριοι και εγκαίρως να ολοκληρώσουμε την ψηφοφορία μας.

Παρακαλώ. Η Επιτροπή Γεωργίας συνεχίζει. Φαντάζομαι χαρήκατε που ήταν τόσο γεμάτη η αίθουσα πριν. Περνάμε λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι στην επόμενη ψηφοφορία. Η είναι ο κύριος Βιέγκας, συντάκτης της γνωμοδότησης, που έχει τον τίτλο «Ο σωστός συνδυασμός χρηματοδότησης για τις περιφέρειες της Ευρώπης. Εξισορρόπηση χρηματοδοτικών μέσων και επιχορηγήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σημαντική γνωμοδότηση, γιατί αφορά τη νέα προσέγγιση που στηρίζει τα χρηματοδοτικά μέσα προκειμένου να τα εξισορροπήσει με τις επιχορηγήσεις στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής. Είναι σημαντικό αυτό για να βρούμε τον σωστό συνδυασμό χρηματοδότησης για τις περιφέρειες και στην επόμενη περίοδο προγραμματισμού. Ποιο θέλει το λόγο, είναι παρόν ο συντάκτης γνωμοδότης, ο κύριος Βιέγκας. Όχι, αλλά είναι παρούσα η συντονίστρια, η κυρία Σένερα. Παρακαλώ. Αν μπορούσαμε να περιμένουμε λίγα λεπτά ακόμα, γιατί νομίζω ότι κάποιο ψάχνει την ε, κάρτα για τι ψηφοφορίε Ο Μιγγέλ έφυγε πιο συγκεκριμένα για να βρει που την έχει αφήσει. Οπότε δύο-τρία λεπτά μπορούμε να τον περιμένουμε ακόμα. <laughs> Μάλιστα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κερδίσαμε χρόνο από την προηγούμενη ψηφοφορία. Οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα περιμένουμε τον uh, κύριο Βιέγας, πολλά δε που είναι και συντάκτης του γνωμοδότησης. Έχω πρόταση. Μια και είναι παρούσα η συγγήτρια της επόμενης γνωμοδότησης, η κυρία Νταντζίλα, ας ψηφίσουμε πρώτα τη δική της γνωμοδότηση. Που αφορά τις συνθήκες εργασίας και την επισφαλή απασχόληση. Όπως είπε η κυρία Βιόριτσα Νταντζίλα είναι η συγγήτρια αρμόδια κατ' ουσίαν επιτροπή είναι Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων και Απασχόλησης. Θα δώσω το λόγο στην εισηγήτρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να σας πω πως ε, Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους και όλους όσους συνεισέφεραν σε αυτή την έκθεση και ελπίζω πως η έκθεση αυτή θα προσφέρει κάποια προστιθέμενη αξία. Να ευχαριστήσω και τη γραμματεία και να σας πω πως όλοι προσπάθησαν πάρα πολύ και νομίζω πως το ζήτημα είναι σημαντικό και επηρεάζει όλους όσους ε, δουλεύουν σε τέτοιες ε, συνθήκες αβεβαιότητας. Σας ευχαριστούμε κυρία Νταντσίλα. Περνάμε στην ψηφοφορία ξεκινάμε με τη συμβαστική τροπολογία Α. Ψηφίζουμε ηλεκτρονικά όπως και πριν τις συμβαστικές τροπολογίες. Άρχεται η ψηφοφορία για τη συμβαστική Α. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 38 της κυρίας Σράιερ. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογία 38. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τροπολογία 39 του κυρίου Καπούτο. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, καλώς. Για την τροπολογία 38 άρχεται ηλεκτρονικός έλεγχος. Λυπάμαι. Αλλά πριν ψηφίσετε υπέρ, κύριε Ταραμπέλα, και η διπλανή. Γι' αυτό θεώρησα ότι υπήρχε πλειοψηφία. Τέλος πάντων, τέλος ψηφοφορίας για την 38. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται όμως γιατί άλλαξαν στάση οι σοσιαλιστές που πριν ψήφιζαν υπέρ. Εν πάση περιπτώσει, τροπολογία 39. Άλλο, άλλη τροπολογία. Άλλο νούμερο ήταν. Ε, δεν πρέπει να κάνουμε λάθο. και νομίζω ότι είχαν πει άλλο νούμερο, άλλον αριθμό δηλαδή τροπολογίας. Α, ah, okay. Okay. Τροπολογία 39. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 40. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 41. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και περνάμε στην τροπολογία 48. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 53 υπέρ. Εγκρίνεται. 55 υπέρ. Εγκρίνεται. 56 υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία σε. Σι. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 59. 59. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 59. Ωραία, εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία Β, α μικρό. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική τροπολογία D. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στις τροπολογίες 71-72. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. 70-71-72. Τώρα περνάμε στις 49. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 82 υπέρ. Εγκρίνεται. 84 υπέρ εγκρίνεται. 74 υπέρ, εγκρίνεται. 75 υπέρ, εγκρίνεται. 77, ποιος είναι υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 78 υπέρ, εγκρίνεται. 79 υπέρ, κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 81 υπέρ. Εγκρίνεται. 86 υπέρ. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 83. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Ισοπαλία. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία F. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στις τροπολογίες 98, 111, 103. Αυτές οι τρεις. Ποιος είναι υπέρ. 98, 101, 103. Εγκρίνονται. Τροπολογία 106. Όχι. 100, εκατό. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. δύο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Ή θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο. Όχι. 104. 104. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 105. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1 από τις αιτιολογικές σκέψεις του κυρίου Νταντά και Σάντερ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 13. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 14. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται λόγω ισοπαλίας. Τροπολογία 18 του κυρίου Ταραμπέλα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Άρχεται η ψηφοφορία για την τροπολογία 18. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 19. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 21. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογίες 22 και 23 μαζί. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνονται. Τροπολογία 24. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 25. Υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 26. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 27. Υπέρ Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 27. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Με μικρή διαφορά. Τροπολογία 28. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 28, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Σας ζητώ συγγνώμη. Ψηφίζουμε την 29. Ποιος είναι υπέρ, υπέρ της 29 εγκρίνεται. Τροπολογία 30, ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης, όπως έχει τροποποιηθεί. Ηλεκτρονικά ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κυρία Νταντσίλα. Μήπως θέλετε το λόγο. Η συγγετρία παρακαλώ. Κυρία Νταντσίλα, μήπως θέλει το λόγο. Ορίστε. Ναι, Δεν θέλετε. Πολύ καλά. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κυρία Νταντσίλα και σας και τους και οδησηγητές, ε, τους συνεργάτες σας. Το, κάνει, <laughs> το έκανε αυτό εκ μέρου μου, κύριο Ταραμπέλα σα ευχαρίστησε ήδη. Τη φιλήσατε κιόλα. Έβγε. Περνάμε στην γνωμοδότηση του κυρίου Βιέγκα. Γνωμοδότηση Βιέγκα. Ήρθε στο μεταξύ ο εισηγητή. Το περιμέναμε. Είπα πόσο σημαντική είναι αυτή η γνωμοδότηση γιατί δημιουργεί ε, νέα προσέγγιση για το σωστό συνδυασμό των χρηματοδοτικών μέσων και των ε, επιχορηγήσεων και στο μέλλον θα έχουμε όλο και περισσότερα τέτοια μέσα και μηχανισμούς και λιγότερες άμεσες ενισχύσεις. Ο κύριος Βιέγκας, ο εισηγητής, θέλει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μία σύντομη παρατήρηση, δεν θέλω να καθυστερήσουμε. Θα ήθελα να επισημάνω το γεγονός ότι καταφέραμε να εκπονήσουμε γνωμοδότηση που θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει σε μεγάλο βαθμό όλο το φάσμα απόψεων της Επιτροπής Γεωργίας. Τα χρηματοδοτικά μέσα ε, λέμε στην γνωμοδότηση ότι είναι ένα εργαλείο με πολλά θετικά σημεία, αλλά τα χρηματοδοτικά μέσα είναι νέοι μηχανισμοί, νέα εργαλεία και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να διακυβεύσουν τις ε, υφιστάμενες πολιτικές στήριξης που ισχύουν για τη Γεωργία και κυρίως στο δεύτερο πυλώνα. Θα πρέπει να εξεταστούν λοιπόν ε, αυτά τα εργαλεία που είναι θετικά, έχουν θετικές πτυχές, αλλά θα πρέπει να εξεταστούν δεόντως και να συνδυαστούν με τα υπόλοιπα μέσα στήριξης της γεωργίας. Όχι με τη λογική της αντικατάστασης, αλλά τη λογική της συμπλήρωσης. Νομίζω ότι αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει η γνωμοδότησή μου, δηλαδή προσοχή και ε, μέρημνα, ώστε να διαφυλάξουμε την παραδοσιακή στήριξη των μέσων ε, του δεύτερου πυλώνα. Είμαι ικανοποιημένο από τη γνωμοδότηση πάντως που επετέφθη χάρη στην αγαστή συνεργασία όλων και της γραμματείας και των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων ευρωβουλευτών με τους βοηθούς τους. Πιστεύω ότι όλοι από κοινού είχαμε πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία. Κάναμε μάλιστα και ακροάσεις, δημόσιες ακροάσεις με εκπροσώπους του γεωργικού κλάδου και έτσι συγκεντρώσαμε μια πλειάδα απόψεων που τροφοδότησαν τη γνωμοδότηση, που θεωρώ ότι είναι ε, συνενετική και ευελπιστώ ότι θα εγκριθεί και με μεγάλη πλειοψηφία. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ τους Πολωνούς ε, διερμηνείς να μιλάνε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο γιατί δεν ακούω καλά πάντα. Ευχαριστούμε τον εισηγητή μας τον κύριο Βιέγκας και περνάμε στην ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία Α, άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και περνάμε στην τροπολογία 39 του κυρίου Ροπέ. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται, σας ευχαριστώ. Τροπολογία 21. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 23. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 79. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 31 του κυρίου Σάνι. Ποιος είναι υπέρ της 31, εγκρίνεται. 32, 33, 34 μαζί. Ποιος είναι υπέρ, εγκρίνεται. 35, υπέρ, κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 35, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία C. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Επαναλαμβάνουμε έναρξη της ψηφοφορίας. Έναρξη ψηφοφορίας για τη συμβαστική τροπολογία C. Ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Δέλτα, D, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 48 του κυρίου Καπούτο. Ποιος είναι υπέρ. Υπέρ τη 48. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία ε. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Περνάμε στην 59. Ναι. Ποιος είναι υπέρ της 59 του κυρίου Νίκολσον. Εγκρίνεται. Τροπολογία 60. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 61 ε, υπέρ. 62 υπέρ. Εγκρίνεται. Και περνάμε στη συμβαστική τροπολογία F, άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την 73, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 75 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 75. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 76. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. 77. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 1. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. εγκρίνεται και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότησης όπως έχει τροποποιηθεί. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συγχαρητήρια κύριε Βιέγας. Μήπως θέλετε το λόγο. Όχι. Συγχαρητήρια και πάλι στον εισηγητή μας και τους συνεργάτες του, τους και ηγητές Και περνάμε στην επόμενη ψηφοφορία, την τελευταία, για το φινικέλαιο. Αρμόδια κατ' ουσία είναι η Επιτροπή Περιβάλλοντος για το θέμα του φινικελαίου και της αποψήλωσης των τροπικών δασών. Εμείς έχουμε γνωμοδότηση, την οποία συνέταξε ο κύριος Μαρτσελέση, που είναι και ο αρμόδιος για να λάβει το λόγο, πιστεύω, ο κατάλληλος άνθρωπος. Παρακαλώ, κύριε Μαρτσελέση, σας ακούμε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω τους και ηγητές για τη συνεργασία τους και φυσικά και τους ε, συνεργάτες μας, ε, τους ε, συμβούλους και κυρίως των Πρασίνων που εργάστηκαν πολύ σκληρά. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω όλους όσους ασχολήθηκαν με το θέμα, γιατί νομίζω ότι αυτό που πετύχαμε είναι ένας μεγάλος βαθμός συνένεσης σε ένα θέμα το οποίο είναι και κοινωνικό και περιβαντολογικό και έχει να κάνει με το πώς η αποψήλωση μπορεί να επηρεάσει, με συγχωρείτε, ένα λεπτό παρακαλώ. Θα ήθελα λοιπόν να τους ευχαριστήσω γιατί το θέμα αυτό της αποψηλώσεις έχει πάρα πολλές ε, επιπτώσεις για θέματα ε, βασικά στην Μαλαισία, στην ε, Ινδονησία και ξέρετε ότι εκεί έχουν αποψηλωθεί δάση. Έκταση ίσως η Γερμανία. Οπότε καταλαβαίνετε πως... Ε, αυτό το είδος ε, ε, ε, ελαιού χρησιμοποιείται είτε για καύσιμα είτε για βρόσιμους σκοπούς στην Ευρώπη. Οπότε το έλαιο φοινικά καταλαβαίνετε ότι στη γνωμοδότηση έτσι όπως το έχουμε τοποθετήσει, ε, λαμβάνει υπόψη και το θέμα της χρήσης χερσαίων εδαφών και τα ανθρώπινα δικαιώματα και θα ήθελα να γνωρίζετε πως η θέση αυτή για το φινικέλο στηρίζεται απόλυτα ή σε πολύ μεγάλο βαθμό από την Επιτροπή και γι' αυτό ευχαριστώ τους συναδέλφους που έκαναν ό,τι μπορούσαν για το θέμα τούτο. Σας ευχαριστούμε κύριε Σιγητά και ευχαριστούμε και τους συνεργάτες. πριν περάσουμε στην ψηφοφορία, θα παρακαλούσε τους συμβούλους των πολιτικών ομάδων να ελέγξουν με τους συντονιστές αν μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα την συνεδρία των συντονιστών που κανονικά έχει προγραμματιστεί για τις 11.30. Ελέγξτε παρακαλώ αν γίνεται, μια και θα τελειώσουμε νωρίτερα τις ψηφοφορίες, να ξεκινήσουμε νωρίτερα και τι συνεδρίες των συντονιστών. Ας το ελέγξουν παρακαλώ οι σύμβουλοι των πολιτικών ομάδων. Και περνάμε τώρα στην ψηφοφορία. Πρώτη συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Συμβαστική τροπολογία 1. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 18. 18. Παρακαλώ, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Τροπολογία 78. Ποιος είναι υπέρ. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 78, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Με μεγάλη διαφορά. Δεν ε, είδα καλά. Συμβαστική τροπολογία 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον εγκρίνεται, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 15. Τέλος. Εγκρίνεται. Περνάμε στην συμβαστική τροπολογία 5, λέει ο Πρόεδρος. Αλλά λάθος, λάθος. Ξεχάσαμε την 131. Ναι. Τροπολογία 139. 131, συγγνώμη, ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 5 τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Περνάμε στην τροπολογία 50. 50. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Τροπολογία 54. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 130. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 119 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία 8. Άρχεται ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 13. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 15. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 16. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία 17. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνατε. Τροπολογία 115. 115. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 112 υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 112. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. Θα ελέγξουμε και την 115. Κανονικά είναι το ίδιο αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 115. Ηλεκτρονικά, παρακαλώ. Τροπολογία 115. Γιατί ίσως είναι το ίδιο αποτέλεσμα με την 112, οπότε καλό είναι να το ελέγξουμε. Τέλος ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και 115. Ζητώ συγγνώμη για πριν. Τροπολογία 170. 170. Ποιος είναι υπέρ. Εγκρίνεται. Και ψηφίζουμε το σύνολο της γνωμοδότης, όπως έχει τροποποιηθεί. Ποιος είναι υπέρ. Άρχεται η ψηφοφορία μάλλον, συγγνώμη, ηλεκτρονικά, ηλεκτρονικά. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται η γνωμοδότηση του κυρίου Μαρτσελέση. Συγχαρητήρια κύριε Σιγητά, δεν ξέρω αν θέλετε πάλι το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε και πάλι, θερμά συγχαρητήρια και ευχαριστούμε και τους ε, σκιώδης ηγητές, βοηθούς κτλ. Ολοκληρώνεται η τακτική συνεδρία της Επιτροπής και αν γίνεται θα ξεκινήσουμε λίγο νωρίτερα τη συνεδρίαση των συντονιστών. Participate.